Ένα βουλευτή βλέπω ότι έχει λησμονήσει την κάρτα ψηφοφορία, αν όμω όλοι οι άλλοι τι έχουν, θα λάβουμε απλώ υπόψη το έξτρα αυτό αριθμό. Έχουμε λοιπόν τώρα το πρώτο θέμα τη σημερινής διατάξεώ μα. Σα υπενθυμίζω ότι οι συνεδρίες των συντονιστών που, προβλέπεται για, το, ως, την αρχή τη σημερινή συνεδριάσεω έχει αναβληθεί για τι 27 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα. Άρα μπορούμε σήμερα να αρχίσουμε αμέσως τη συνεδρίαση και να την ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρία στις 12.30 χωρίς να έχει αυτό καμιά επίπτωση στο, στην απογευματινή. Στις 3 η ώρα θα αρχίσουμε με την ομιλία του Έλληνος Υπουργού Γεωργίας. Η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Αν δεν έχετε ενστάσεις για τα πρακτικά τα θεωρώ εγκεκριμένα. Και έρχομαι στον αριθμό 4 της ημερησίας διατάξεως. για την διαχείριση των δαπανών στην αλυσίδα τροφίμων, προστασία της υγείας και, της, ε, και γενικότητα των ζώων, επίσης για προϊόντα αναπαραγωγής φυτών με ναι, εισηγήτρια την κυρία Λεμπρό η οποία θα εξηγήσει τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου και το ενοποιημένο κείμενο και έχουμε και την έκθεση για τα τρόφιμα και καθώς και για τις ζωοτροφές και βλέπω στις προφορίες που έχω ενώπιον μου ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία. Μόλις μου λένε ότι αναβλήθηκε το θέμα. Και τότε λοιπόν προχωρούμε στην ψηφοφορία. Επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να σας εξηγήσω. Ο Πρόεδρος. Καλά. Προχωρούμε στο θέμα 5 της ημερησίας διατάξεως. Το μέλλον του τομέα ποροκυπευτικών στην Ευρώπη. Στρατηγικές για ανάπτυξη. Πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, την οποία καλούμεθα να ψηφίσουμε. Έχουμε 167 τροπολογίες, υπάρχουν ήδη συμβιβαστικέ τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και αυτό βεβαίως διευκολύνει την ψηφοφορία. Επιθυμεί να λάβει το λόγο μήπως η συγγήτρια. Εφόσον με προσκαλείτε να λάβω το λόγο, ε, δέχομαι κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Μάκιντάιρ. Πρόκειται για την πρώτη μου έκθεση στην ε, παρούσα επιτροπή και είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων για την συνεργασία που μου προσφέρθηκε. Όπως είπατε είχαμε 167 τροπολογίες. Καταβάλαμε λοιπόν σημαντική προσπάθεια για να μειώσουμε τον όγκο της λίστας ψηφοφορίας και Επαναλαμβάνω, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από την διάθεση συνεργασίας που διαπίστωσα από όλε τις πολιτικές ομάδες και ελπίζω ότι καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορέσει να ε, γίνει δεχτό από όλες τις πλευρές στην ε, Επιτροπή μας. Είναι γνωστό πόσο σημαντικά είναι τα οποροκυπευτικά και κυρίως σαν ποσοστό της συνολικής αγροτικής παραγωγής που απασχολεί και τόσο περιορισμένο έδαφος έκταση. Ελπίζω, παραλαμβάνω, ότι θα ε, τύχει μεγάλη υποστήριξη σήμερα και επαναλαμβάνω τις ευχαριστήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία εισηγήτρια. Προχωρούμε στην ε, ψηφοφορία. Συμβαστική υπαριθμόν 1. Ποιος είναι υπέρ. Παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι. Απλώς. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική ήττα ή age. Α, για την 40 ζητείτε πρώτα ηλεκτρονική επαλήθευση που την ανοίγω τώρα. Λήξη. Εγκρίνεται 31 προς 20. Η συμβαστική ήττα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική Ι ή I. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ε, τώρα η 53. Ψηφίζουμε την τροπολογία 53. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ας γίνει καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Λήξεις. Εγκρίνεται. Η επόμενη τροπολογία είναι υπαριθμών 54 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η συμβαστική J υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Έχουμε ακόμα την 55 πρώτα συμβαστική, 55, ε, συγγνώμη, τροπολογία 55 υπέρ. Μάλιστα θα κάνουμε αμέσως και επαλήθευση. Να με συγχωρείτε πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Ελήξη. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Συμβαστική J. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Υπαριθμών 62 υπέρ, κατά, επαλήθευση, αρχίζει, λήξη, πρόκειται για ισοψηφία αν καταλάβαμε καλά. 17 υπέρ, 17 κατά, άρα απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, ούτε και εδώ είναι το αποτέλεσμα απόλυτα σαφές. Θα επαληθεύσουμε λοιπόν. 63 αρχίζει. Τέλος. Απερίφθη. 64. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Αρχίζει. εγκρίνεται Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα Όπως έλεγα λοιπόν, συμβαστική κάπα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69 της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λάμδα υπέρ. Λάμδα ή L υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Με μία ψήφο κατά. Ακολουθεί η ελ υπερ κατα εγκρινεται και αυτη με μια ψηφοκατά ακολουθει η υπαριθμον 75 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξεις. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Καλά λοιπόν που κάναμε και την επαληθεύση. Είναι 17 προς 16, αλλά ο κύριος Λάιν που έχει ξεχάσει την κάρτα του ήταν κατά. Τώρα η συμβαστική μη. Ε, μ ή μη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. μόνο 85. Υπέρ. Κατά. Μου φαίνεται ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Όντως εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία νη, όπως Νοέμβριος, αρχίζει η ψηφοφορία. ψηφιπέρ μάλλον, ψήφι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται αυτή. Τροπολογία 89. Υπέρ. 89, ε. ευχαριστώ. Κατά. Ας κάνουμε παρήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξεις. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Λέω πρόεδρο 91. Α, όχι, πράγματι. 90 είναι το σωστό, όπως μου λέει η γραμματεία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά απορρίπτεται 93 υπέρ κατά απορρίπτεται 94 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή συμβαστική όμικρον υπέρ Εγκρίνεται. 97 του κ. Χόισλινγκ υπέρ. Και τώρα λαϊκό κόμμα είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. κατά. Εγκρίνεται ή μήπως προτιμάτε να γίνει επαλήθευση. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν για την 97 λήξης. Εγκρίθηκε όντως. Η συμβαστική π υπέρ κατά εγκρίνεται και ακολουθεί η συμβαστική Q υπέρ, κατά. Εγκρίνεται και αυτή η συμβαστική τροπολογία. 102 δεκάστρο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξεις. Λήξεις όπως είπα έληξε η ψηφοφορία και απερίφθη η τροπολογία. Συμβαστική R ή ρο υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική S σίγμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβαστική ταφ υπέρ κατά εγκρίνεται. Παρακαλώ, ε, συμβαστική γιου υπέρ κατά εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά εγκρίνεται. 125 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Κατά. Εγκρίνεται. 126 υπέρ. 126 κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μία επαλήθευση. Παρακαλώ. Zamykam głosowanie. Teraz. 126. 19 προς 14. Εγκρίνεται. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Όχι. Συμβαστική Β. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Εγκρίνεται. 131. Υπέρ. Κατά. απαραίτητα. Ε, w. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική X. Υπέρ. Υπέρ. Κύριε Ντες. Α, εντάξει, ψηφίσατε. Εγκρίνεται. Συμβαστική, ή μάλλον τροπολογία 140 του κυρίου Ντάντα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική Y, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά εγκρίνεται 147 υπέρ κατά εγκρίνεται τώρα η τροπολογία ΑΣ υπέρ κατά εγκρίνεται και ακολουθεί η 150 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 155 του κ. Ντεκάστρο, αλλά δεν φαίνεται να είναι σωστό. 152 λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά εγκρίνεται του κ. και 153 υπέρ κατά. αλλά θα επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα η συμβαστική Ζήτα υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται ωστόσο προτιμώ να επαληθεύσουμε αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία για την ζήτα λήξεις Και συνεχίζουμε. Τροπολογία 156. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 156. Λήξη. απορρίπτεται. 157 υπέρ. Ναι, λέει ο πρόεδρος, λάθος, είπα 159 υπέρ. Υπέρ, κατά, Εκατόν εξήντα ένα υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΑ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 164 Νικουλέσκου υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τέλος ευχαριστώ πολύ απορρίφθηκε Εκατόν εξήντα πέντε. υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΒ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Και τώρα οι αιτιολογικές σκέψεις, οι εκτιμώντας, υπαριθμόν ένα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. δύο, υπέρ, εγκρίνεται. τρία, υπέρ, εγκρίνεται. τέσσερα, υπέρ, Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξεις. απεριφθιόντως 5 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Η συμβαστική σε υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται και αυτή. Υπαριθμόν 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Ψηφίζουμε τη 17. Κατά τώρα. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξεις. εγκρίνεται. 17 του κύριου Χόισλινγκ. Υπέρ. Εγκρίνεται. Ο πρόεδρος αυτοδιορθώνεται λέγοντας ότι τη 17 την έχουμε ήδη ψηφίσει. Και σωστό είναι. 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και ακολουθεί η, παριθμόν, η συμβαστική ε, μάλλον F. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. Και τώρα η παριθμόν 24 υπέρ. 24 κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αυτή απορρίπτεται ή πιστεύετε ότι πρέπει να επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία για την 25 λήξη Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 30. Δεκάστρο. Υπέρ. και σε επαληθεύσουμε καλύτερα το αποτέλεσμα, κάνοντας ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μου φάνηκε ότι ήταν σαφές, αλλά τελικά δεν είναι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την, 10, για την 30 μάλλον, έδειξε τώρα. Εγκρίνεται. 31 Χόισλινγκ υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Αρχίζει. λίγοι Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Ας γίνει και εδώ επαλήθευση καλύτερα που αρχίζει τώρα για την 33. Έληξε. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά αποχές. Όχι αποχές δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Ψήφι υπέρ επαναλαμβάνω. Όχι, θα γίνει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία αυτή. Αρχίζει λοιπόν τώρα. Έληξε. Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο. Και Λάιον, είστε υπέρ Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ακολουθεί τώρα η ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Πόλσεν. Έχουν κατατεθεί 104 τροπολογίες, 9 συμβιβαστικές έχουν προταθεί από τις πολιτικές ομάδες. Κυρία Πόλσεν θέλετε το λόγο πριν την ψηφοφορία. Так, Pre-posted, though. Pre-posted, tak? To jest to? Proszę Państwa, otwieram, otwieram głosowania. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ δεκτή. Δύο. Ευχαριστώ δεκτή. Τρία. Ευχαριστώ δεκτή. Τέσσερα. Δεκτή. Πέντε υπέρ. Ευχαριστώ δεκτή. Έξι υπέρ. Δεκτή. Tak, amendment, poprawka 22. To jest za poprawką 22. 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Είκοσι τρία υπέρ. Κατά. Δεκτή. Είκοσι τέσσερα υπέρ. Δεκτή. 25. Α, για μια στιγμή. «27». 27 θα ψηφίσουμε την 27. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως για την 28 ψηφίζουμε. Α, όχι, δεν ψηφίζουμε. Θα περάσουμε στις 29. Ποιοι είναι υπέρ. Ε, ζητώ συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Ο κύριος Μποβέ ε, ήθελε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά μετά μετάνιωσε. Οπότε αναγκάστηκα και εγώ να μετανιώσω, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, 29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 31. Ποιοι είναι υπέρ της 31. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Ο κύριος Λάιον είναι υπέρ. Έτσι και αλλιώς απορρίπτεται. 16 υπέρ, 16 κατά. Α, όχι. Ναι, όχι. Τελικά απορρίπτεται. Εν πάση περιπτώσει επανέρχεται ο πρόεδρος. Απερίφθη. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική υπαριθμών 1. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 35. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική υπαριθμών 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ δεκτή. Περνάμε τώρα στην 40. Ποιοι είναι υπέρ της 40. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. 45. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 4. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 45. Επανέρχομαι στη 45 και ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Απερίφθη. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ τη συμβιβαστικής 4. Ευχαριστώ. Δεκτή. 48 ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Απερίφθη. Περνάμε στην 49. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ δεκτή. 47 υπέρ του κυρίου Λάιον. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 52. Υπέρ. Ευχαριστώ. 53 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 54 υπέρ δεκτή. 82 υπέρ. Έχει καταπέσει, συγγνώμη. Συμβιβαστική 6, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ, δεκτή. 7, ποιοι είναι υπέρ της 7, δεκτή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Θέλετε να γίνει έλεγχος. Θα ελέγξουμε συνεπώς για την 65. Τέλος. Κύριε Λάιον, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Δεκτή. 70. Ποιοι είναι υπέρ της 70. Δεκτή. 71 υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ της 71. Ποιοι είναι κατά. Κατά. Δεκτή. 72. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ελέγχουμε την 71. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκαεπτά υπέρ, 17 κατά, συνεπώς απορρίπτεται. Τροπολογία 72. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ τη συμβιβαστική 9. Δεκτή. 80. Ποιοι είναι υπέρ τη 80. Ευχαριστώ. έχει καλυφθεί η 80 από άλλη τροπολογία και γι' αυτό περνάμε στην 81 αμέσως. Ποιοι είναι υπέρ της 81. Δεκτή. 83 υπέρ. Έχει καταπέσει και η 83. 84. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. 86. Ποιοι είναι υπέρ της 86. Κατά. Δεκτή. Συνεπώς περνάμε στην 90. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 91. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 93. Έχει καταπέσει. 94. Ποιοι είναι υπέρ της 94. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή.

Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Απερίφθη. 99. Κατέπεσε. Όχι, δεν κατέπεσε. Ψηφίζουμε την 99. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην εκατό. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Εκατόν ένα. Υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απερίφθη. Εκατόν δύο, Ποιοι είναι υπέρ. Εκατόν τρία. Ή όχι, εκατόν τέσσερα. Επανέρχεται ο πρόεδρος. Εκατόν τέσσερα υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα θα περάσουμε στην 7. Ποιοι είναι υπέρ δεκτό. Οκτώ. Ευχαριστώ. Δεκτή. 9. Ποιοι είναι υπέρ. 9. Κατά. Δεκτή. 10. 10. Ποιοι είναι υπέρ της 10. Δεκτή. 11. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 12 υπέρ. κατά δεκτή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεκατέσσερα υπέρ. Δεκτή. Δεκαπέντε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 16. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται. 17. Ποιοι είναι υπέρ. 18. λάιον Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 19 υπέρ. 19 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ή θέλετε να γίνει έλεγχος. Θα ελέγξουμε λοιπόν για την 19. Τέλος. 14 υπέρ 16 κατά. Ναι, απερίφθη. Poprawka, poprawka 20, 20. Poprawka. 20. Α, 20 ψηφίζουμε λοιπόν. Κατά. 21 μάλλον. Ποιοι είναι υπέρ της 21. Κατά. Απορρίπτεται. το σύνολο του κειμένου όπως το η Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Κύριε Λάιον. Κάτι θέλετε. Θα περάσουμε στο 7 τώρα. γνωμοδότηση Ράιμερ. Εφαρμογή κανόνων και νομικών ρυθμίσεων. Η υπεύθυνη επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και υπάρχουν μοιρασμένε αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 50 για συγκεκριμένα άρθρα. 398 τροπολογίες έχουν κατατεθεί, έχουν όμως προταθεί και 9 ομαδικές ψήφοι. Λοιπόν, ξεκινάμε εκτός αν η κυρία Ράιμερς θα ήθελε το λόγο. Αν θέλετε έχετε το λόγο κυρία Ράιμερς. Όχι, δεν το επιθυμεί η κυρία Ράιμερς. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Πρώτη ομαδική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Κατά επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρώτη ομαδική ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 15 υπέρ 15 κατά απερίφθη. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τη δεύτερη ομαδική ψήφο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την ομαδική 2. Τέλος. Απερίφθη, είναι σαφές. Περνάμε τώρα στην 24. Ποιοι είναι υπέρ της 24. Ποιοι είναι κατά της 24. Απορρίπτεται. 96. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Δεκτή. 28 δεν θα ψηφίσουμε. 101 υπέρ. Δεκτή. 102 θα επαναλάβουμε την τελευταία ψηφοφορία. Για την 102 προφανώς εννοεί ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν κατάλαβε. Εγώ δεν άκουσα να μου ζητήσετε να ψηφίσω για την 102, άκουσα απλά ότι έγινε δεκτή. που να φτάσει η μετάφραση σε μένα είχε περάσει η ώρα. Κοιτάξτε, ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Όταν βλέπω ότι οι συντονιστές ε, εκφράζονται ομόφωνα υπέρ μιας τροπολογίας, δεν ζητώ ε, ε, ποιοι είναι κατά να μάθω γιατί βλέπω ότι είναι διαμορφωμένη η ψηφοφορία. Τυπικά δεν είμαι εντάξει βέβαια αλλά πάω γρήγορα. Λοιπόν από εδώ και πέρα θα είμαι πιο προσεκτικός. Κοιτάξτε, το, το κατανοώ αυτό που είπατε, αλλά εγώ δεν άκουσα καν ότι ζητήσατε να μας ψηφίσουν. Θα φταίει η ερμηνεία βέβαια. εντάξει, ε, συνεχίζουμε με την 101 εκ νέου, 101 ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 101. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 102. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 105. 105 παρακαλώ. Όχι, όχι, αφήστε τη αυτή. 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 106. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 107. Υπέρ. κατά απορρίπτεται 35 υπέρ κατά δεκτή εκατόν δέκα ποιοι είναι υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 110. Τέλος. Απορρίπτεται. 112. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 36 υπέρ. Δεκτή. 114 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την 114. Τέλος. Απορρίπτεται. 116. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 118. Τέλος. Δεκτή. 119. 120. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 121. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 37. Υπέρ. Δεκτή. 38. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Υπαριθμού 40. Oh, yes. Okay, 125. Καλά, 145. 125. Λιπέρ. Κατά. Όχι. Απορρίπτεται. Τώρα η 40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 128 υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σαράντα ένα. Σαράντα ένα. Υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. 135. Θα ψηφίσουμε για την 135. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά εγκρίνεται 140 υπέρ κατά εγκρίνεται 100 όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 42, υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 142 τώρα. Υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνατε. 143 υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 143. Πέρες ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Κύριε Λάιον. Τώρα θα περάσουμε στην 145 υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 100. Διόρθωνα, ο πρόεδρος. Η τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 44 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά απορρίπτεται 45 υπέρ Ευχαριστώ κατά. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Ευχαριστώ εγκρίνεται. 151. Πάλι τη ηγέτρια μου υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 152. 152. Υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Εγκρίνεται. 153. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 155. Κατά. Εγκρίνεται. 156. Υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 47. 47. Υπέρ, εγκρίνεται. 147. Διαδικαστικό από την εισηγήτρια. ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ελευθερία εντολής. Δεν αρκεί να κοιτάτε τους συντονιστές. Κάθε βουλευτής μπορεί να έχει και διαφορετική άποψη. Και πρέπει καταρχήν να ρωτάτε υπέρ, κατά, αποχές. Ε, δέχομαι αυτό το σχόλιο. Τροπολογία 47 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 157. Ε, Υπέρ. Όχι, ζητά συγγνώμη, πρόεδρο, διορθώνει την 48 θα ψηφίσουμε, αλλά την έχει αποσύρει ήδη η συγγήτρια.

Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Απορρίπτωτα. 164. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτωτα. Θα κάνουμε μία επαλήθευση. Για την 164, παρακαλώ. Πανιέ. Πέρας. Απορρίπτεται. Απερίφθη 164-49 υπέρ 49. Κατά. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά εγκρίθηκε 166 υπέρ κατά εγκρίνεται η 50 της εισηγητρίας υπέρ ευχαριστώ κατά εγκρίνεται 51 της εισηγήτριας και πάλι υπέρ κατά εγκρίνεται 168 όχι δεν θα την ψηφίσουμε 52 της εισηγήτριας 52 υπέρ κατά εγκρίνεται 169 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 172 είπε. Κατά. Yeah. Θα κάνουμε επαλήθευση. 172. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 174. Kto jest za poprawką 174? 174. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 175 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. το. 178 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. 182. Κατά. Επαλήθευση ηλεκτρονική για την 182. Πέρας. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εντάξει, επαλήθευση για την 186. 186 ψηφίστε παρακαλώ. 186. Απερίφθη. 187. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 87. Πέρες. Απορρίπτεται. Τώρα, ε, μπλοκ ε, ψηφοφορία ε, συνολική, υπαριθμού 4, υπέρ, κατά, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε και μία επαλήθευση. Ψηφίστε. 53 ε, υπέρ. Όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε τώρα για την, ε, ε, για την ομάδα 4, block vote 4, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Εκατόν Όχι, θα γίνει επαλήθευση. Πάλι για την ε, ε, ε, ε, ε ψηφοφορία 4. Το βάνια. Υπέρ, κατά. Μάλλον ψηφίστε ηλεκτρονικά. Τα κούπα του czwarty. Ποπράβκα 189 τα takim Το είναι ζα ποπράβκο 189. 189. Απορρίπτεται 189. Κατά. Απορρίψτε. 190 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται.

Όχι, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. 199. 199. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 201. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Για την 201 παρακαλώ. Zamykam Πέρας. Δεν Απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά απορρίπτεται. 203 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται. 204 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Θα κάνουμε μια επαλήθευση. Zamykam głosowanie, przepraszam. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 205. 205. Όχι, επανερχόμεθα στην 202. Ψηφίζουμε για την 202 ηλεκτρονικά. Τέλος. Τέλος. Απερίφθη. 203 ψηφίζουμε. 203 ηλεκτρονικά. Τέλος. Δεκτή. 205. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 207. Ποιοι είναι υπέρ της 207. Κατά. Απερίφθη. 208. Κατά. Απερίφθη. 59. Όχι, συγγνώμη, το το πρόεδρος 210 υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. 213 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15. 215 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 217 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62. Όχι, συγγνώμη. 219 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 219. Άλλωστε είναι και δική μου τροπολογία, λέει ο κύριος Γεκεύσκη. Τέλος. Απερίφθη. 220. 220. ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 221 ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για την 221 τέλος είχε γίνει τελικά δεκτή. Η 222 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 228, 228 τώρα λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 229 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 229. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή πέντε υπέρ κατά δεκτή. Διακόσια τριάντα υπέρ. Κατά. Δεκτή. Διακόσια εικοσιένα υπέρ κατά δεκτή 232 δεκτή 236 ποιοι είναι υπέρ κατά ποιοι είναι κατά της 236 ηλεκτρονικός έλεγχος Τέλος. 25 przyjęta. Ποπράφκα 237. Kto είναι ζα. Δεκτή. 2.37 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 67. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 2.38 υπέρ κατά δεκτή 2.39 υπέρ κατά απορρίπτεται 240 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Α, επανέρχομαι, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 242. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 243. Ψηφίζουμε. Α, για μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Sprawozdawcy. Kto jest 68 sprawozdawcy. jest za? 68 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 244 υπέρ. Α, για μια στιγμή. 69 ψηφίζουμε τώρα. Την 69 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 70 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ομάδα τροπολογιών 5. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 245. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 246. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 248. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 248. Τέλος. Απερίφθη. 249. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 251. Ποιοι είναι υπέρ. 251 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 252. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 2.53. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Η 2.53 λοιπόν ήταν αυτή, έγινε δεκτή. Α, θα επαναληφθεί όμως η ψηφοφορία για την 2.53. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Τέλος. Έκανα κάποιο λάθος, λέει ο πρόεδρος. Γίνεται δεκτή, περνάμε στην 2.55, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 56. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 257 ψηφίζουμε. Τέλος. 16 υπέρ, 14 κατά γίνεται δεκτή. 2.59 υπέρ. Κατά. κατά, απορρίπτεται. 262 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 263 υπέρ. Υπέρ, κατά, ποιοι είναι κατά, απορρίπτεται. 264 Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. 2.65. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 266 ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 267 ποιοι είναι υπέρ, κατά, Δεκτή. Πηγαίνουμε στην έκτη ομαδική. Είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την ομαδική 6. Τέλος. Δεκτή. Συνεχίζουμε με την 2.72. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 2.73. Ποιοι είναι υπέρ της 2.73. Κατά. Απορρίπτεται. 2.74. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. 2.75. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 276 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος Ψηφίζουμε για την 277. Τέλος. Δεκτή. Με μεγάλη πλειοψηφία. 78. 278. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 279 2, 7, 9, υπέρ κατά δεκτή 280 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 281 υπέρ κατά απορρίπτεται 282 ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 283 υπέρ κατά απορρίπτεται 284 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 78 υπέρ κατά δεκτή 285 υπέρ κατά απορρίπτεται 286 υπέρ κατά δεκτή 287 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 288 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 289 υπέρ κατά δεκτή 290 υπέρ κατά δεκτή 291 υπέρ κατά δεκτή 292 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 292. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 2.93 υπέρ. Κατά. δεκτή. 2.94 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 2.95 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην ομαδική 7. Ποιοι είναι υπέρ της 7. Κατά της ομαδικής 7. Δεκτή. Πάμε στην 300. Ποιοι είναι υπέρ της 300. Κατά. απερίφθη. Αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 300 τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 301. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 303 και είναι υπέρ κατά ελέγχουμε την 303 ηλεκτρονικά Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. έχω κάποια προβλήματα, έχω μια μικρή σύγχυση εδώ. Πάντως είμαστε στην 302. Σηκώστε παρακαλώ τα χέρια σας κατά 304. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα τεχνικά. Η συγγήτρια. παρακαλώ όταν λέτε πάρα πολλά πράγματα μαζί να τα λέτε λίγο πιο αργά γιατί η διερμηνία στα γερμανικά καθυστερεί. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θα προσπαθήσω. 302 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά εγκρίνεται αλλά θα επαληθεύσουμε την 304 αρχίζει η ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία για την 304 έληξε τώρα απορρίπτεται 305 υπέρ όχι λέει ο πρόεδρος 307 υπέρ κατά εγκρίνεται 308 υπέρ κατά εγκρίνεται 310 υπέρ όχι, δεν ψηφίζεται αυτό, συγγνώμη. 309. 309 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, όχι, θα επαληθεύσουμε την 309. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Έληξε. Απερίφθη. 85 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, θα υπαλληθεύσουμε την 85. Αρχίζει. Έληξε. Απερίφθη. 313. Ψηφί υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 314 υπέρ απερίφθη. 315 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή. 316 υπέρ κατά εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και ακολουθεί 318 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Και επαναλαμβάνω, μάλλον επαληθεύουμε την 319 όπου αρχίζει η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. 320. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 321. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 322. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 323. Υπέρ κατά επαληθεύουμε 323 αρχίζει η ψηφοφορία λήξη απερίφθη 324 υπέρ κατά απορρίπτεται. 325 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 326 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 327 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3.28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 329 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 330 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. Ακολουθεί το, η συνολική ψηφοφορία, μπλοκ δηλαδή, υπάρχει μόνο 8 ψήφι υπέρ. Κατά, αλλά ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απερίφθησαν. Και συνεχίζουμε με την 338 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Το μπλοκ τώρα υπαριθμών 9. ψήφι υπέρ αυτού του συνόλου τροπολογιών κατά εγκρίνονται όμως μια στιγμή ο κύριος Ντες ζήτη επαλήθευση αρχίζει για το 9 λοιπόν μπλοκ παριθμών 9 έληξε Απερίφθη. 342 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 343 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 344 υπέρ κατά εγκρίνεται 345 υπέρ κατά απορρίπτεται 346 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή 347 της κυρίας Αγιούσου υπέρ... ...κατά Εγκρίνεται. 348 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 349 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 350 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 351 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 352 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 353 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 354 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 355 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 356 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή. 357 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 358 υπέρ εγκρίνεται 359 υπέρ κατά εγκρίνεται 360 υπέρ κατά απορρίπτεται 361 υπέρ κατά εγκρίνεται 362 υπέρ κατά εγκρίνεται 363 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. 364 υπέρ. 364 κατά. Απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 366 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 367 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 368 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 369 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 370 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 371 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πρώτα θα επαληθεύσουμε την 371. Αρχίζει η ψηφοφορία.

απορρίπτεται 375 υπέρ κατά εγκρίνεται ζητείτε επαλήθευση καλά λοιπόν επαλήθευση 375 τέλος εγκρίνεται 376 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 377 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή. 378 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 379 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 380 υπέρ κατά ας κάνουμε επαλήθευση 380 αρχίζει η ψηφοφορία έληξε εγκρίνεται με διαφορά τεσσάρων ψήφων 381 υπέρ κατά απορρίπτεται 382 υπέρ κατά απορρίπτεται επαλήθευση 382 αρχίζει η ψηφοφορία έληξε απορρίπτεται 383. 383 υπέρ. Κατά. Και αυτό θα επαληθευτεί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται με διαφορά τεσσάρων ψήφων. Και αρχίζει η ψηφοφορία της τροπολογίας 86 ψήφι υπέρ. Υπέρ, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και ακολουθεί 91. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Και μένει πλέον η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως όπως τροποποιήθηκε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Έληξε. εγκρίνεται η γνωμοδότηση και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Przerwa, proszę Państwa, spotykamy się o godzinie 15 z Panem Ministrem. Κυρίες και κύριοι, θα συναντηθούμε στις 3 το απόγευμα και θα συναντήσουμε στις 3 το απόγευμα τον Έλληνα Υπουργό που εκπροσωπεί την ε, Προεδρία. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε όμως και το θέμα υπαριθμό. Α, όχι, όχι, δεν θα συναντηθούμε στις τρεις. Ε, έχουμε και άλλο ένα θέμα. Bo później koordynatorów nie ma. Chciałbym złożyć sprawozdanie z Έχουμε ένα άλλο θέμα λοιπόν στην περισσία διάταξη. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων στην περιοχή της Ριόχα. Εγώ ήμουν επικεφαλής της συγκεκριμένης αντιπροσωπείας. Και θα ήθελα να παρουσιάσω το τι συνέβη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής πήγαμε στην Ισπανία από τις 28 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για οργανωτικούς λόγους. Δεν μπορέσαμε να σας ενημερώσουμε νωρίτερα και είμαι ιδιαιτέρως ευχαριστημένος που είμαι σε θέση να το κάνω τώρα. Να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Χεράν Σκαρθία διότι οργάνωσε πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη επίσκεψη και την παραμονή μας γενικότερα εκεί. Το πρόγραμμα είχε σαν στόχο ε, την γεωργική παραγωγή φυσικά, την μεγάλη σημασία που έχει στην περιοχή της Ριόχα ο αμπελοϊνικός τομέας, αλλά ασχοληθήκαμε και με τα οποροκυπευτικά όπως και με τη τυροκομεία. Είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις, μάθαμε πολλά σχετικά με τα θέματα διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγής Υπήρχε μαζί μας η κυρία Λούλινγκ η οποία είναι και πρόεδρος στο Intergroup για το κρασί στο Κοινοβούλιο. Ήταν μαζί μας και ο κύριος Καπούλας Σάντος όπως επίσης και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Στο πρόγραμμά μας είχαμε συνάντηση επίσης και με τον Ισπανό Υπουργό Γεωργίας, τον πρόεδρο της αυτόνομης κοινότητας της Ριόχα, συναντηθήκαμε με οργανώσεις των γεωργών και με το τοπικό συμβούλιο που ελέγχει τη ονομασία προέλευσης των κρασιών της περιοχής. Επισκεφθήκαμε και ένα τυροκομείο και επισκεφθήκαμε φυσικά και την μπελοϊνική ε, περιοχή μια εξαιρετικά όμορφη περιοχή της Ισπανίας. Ήταν μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Είδαμε τους εξαιρετικούς τρόπους προώθησης των γεωργικών προϊόντων, είδαμε την συνεργασία των γεωργών με τις τοπικές αρχές. Είναι αλήθεια ότι οι περιφερειακές αρχές αφιερώνουν τεράστιες προσπάθειες στην στήριξη των τοπικών παραγωγών κρασιών και τυριών στη Ριόχα. Μιλήσαμε για τα θέματα της ποιότητας, της προώθησης των προϊόντων αυτών που είναι πασίγνωστα σε όλο τον κόσμο. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πόσο ε, ισχυρή είναι η υποστήριξη των τοπικών αρχών της γεωργίας της παραγωγής, κρασιού, τυριού και όλου του τομέα. Υποστηρίζουν επίσης και ε, την παραγωγή αλλά και την πρόθεση των προϊόντων. Ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για άλλες χώρες και για άλλες περιοχές. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Χέραντς Γκαρσία για την εξαιρετική οργάνωση της συγκεκριμένης επίσκεψης. Δεν ξέρω αν θα ήθελε το λόγο η κυρία Χέρανς Γαρσία. Έχετε τη δυνατότητα αυτή και το προσωπικό σας βοήθησε στην οργάνωση της επίσκεψης. Παρακαλώ κυρία Γκαρσία να μεταφέρετε τα ευχαριστήριά μας στο προσωπικό του γραφείου σας και στις περιφερειακές αρχές. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ήθελα μόνο να επιβεβαιώσω αυτά που μας είπατε μόλις και να σας συγχαρώ διότι γηθήκατε της αποστολής με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Ε, νομίζω ότι λίγες ε, περιοχές ε, μπορούν να είναι περήφανες για ένα τόσο ζωντανό γεωργικό τομέα. Οι αρχές και ο πληθυσμός είναι προσιλωμένοι στην γεωργία και κυρίως στην αμπελουργία ε, και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, πολύ καλά οργανωμένη. Ε, μας επιφύλαξαν πάρα πολύ καλή υποδοχή οι Ισπανικές αρχές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Εστέρ για την ε, επίσκεψη που οργάνωσε και τον αντιπρόεδρο που ηγήθηκε της αποστολή αυτής με τόσο αποτελεσματικό τρόπο. Ε, Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Η κυρία Χέρι Γκαρσία θα πάρει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστούμε και πάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Σεκεύσκη. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Καπούλα Σάντος για τα καλά του λόγια να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, της ε, Επιτροπής που επισκέφθησαν τη Ριόχα, την περιοχή μου. Είναι γνωστός ο στόχος της επίσκεψης αυτής, να γνωρίσουν δηλαδή μια γεωργική πραγματικότητα, μια γεωργική κυρίως περιοχή, κτηνοτροφική επίσης, και με μια βιομηχανία η οποία συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Έκανε εντύπωση η επίσκεψη αυτή στην περιφέρειά μου. Επίσης ε, και η παρουσία του Μιγουέλ Άριας, του Υπουργού, όπως επίσης και του Προέδρου της Περιφερειακής Κυβέρνησης και των Συμβούλων του Τοπικού Κοινοβουλίου έκανε έτσι ώστε, έκαναν έτσι ώστε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά, τα περιφερειακά αλλά και τα εθνικά να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στη Ριόχα, κάτι το οποίο λοιπόν απασχόλησε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στις γειτονικές περιοχές. Υπήρξε λοιπόν ενδιαφέρον, ήταν επιτυχής η επίσκεψη είναι ιδιαίτερα ευτυχής η τοπική παραγωγή που μπόρεσαν με κάθε ειλικρίνεια να ομιλήσουν άμεσα, να συνομιλήσουν άμεσα με τους ευρωβουλευτές. Προσπαθούν να εκφραστούν συνήθως και να προωθήσουν τα θέματα τους μέσω των εθνικών εκπροσώπων τους και θέλει και η περιφερειακή κυβέρνηση να ευχαριστήσει για τα καλά λόγια που είπατε για την περιφέρεια και την παραγωγή της περιφέρειας και εγώ θα ήθελα επίσης όταν επισκεφθήκαμε de Εν πάση περιπτώσει τα θέματα των κτηνοτροφικών μονάδων που αποτελούν σημαντικά σημεία ανησυχίας για την περιοχή και είδαμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον με πόσο σωστό τρόπο χρησιμοποιήθηκαν τα, τα χρήματα του ΦΕΝΤΕΡ και για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και για την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ενέργειας και των υδάτινων πόρων κτλ. Ε, είδαμε λοιπόν και την πραγματικότητα που ισχύει στην περιοχή στην Ριόχα ε, Μπάχα, είναι μια μικρή, στην κάτω Ριόχα είναι μια πάρα πολύ ε, μικρή περιοχή, εντελώς διαφορετική από την Άνω Ριόχα και την πρωτεύουσα της περιοχής, οι συνθήκες, ε, οι οικονομικές, γεωργικές είναι εντελώς διαφορετικές και τις γνωρίσαμε. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στις τοπικές αρχές. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε εσάς και τους βοηθούς σας. Ήταν πάρα πολύ καλή οργάνωση της αποστολής. Για την Γεωργία Μικρής Κλίμακος εγώ ήμουν ο εισηγητής και ομολογώ ότι έμαθα πάρα πολλά. Ε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης για τον ε, αμπελίνικο τομέα. Ήξερα ότι είναι καλά οργανωμένος, αλλά ο γαλακτοκομικός ε, τομέας ήταν αυτός που με εντυπωσίασε. παραγωγή, μικρή παραγωγή, που έχουν κατσίκες, πρόβατα. και εργάζονται ε, με πάρα πολύ αποτελεσματικό, συνεργάζονται ε, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο με την μεταποιητική βιομηχανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στη δική μου τη χώρα, την Πολωνία. Οι μικροί παραγωγοί χρειάζονται την υποστήριξη των τοπικών αρχών, ούτω ώστε να εξασφαλίσουν ε, τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Χρειαζόμαστε ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο για να βελτιωθεί η παραγωγή των μικρών μονάδων. Στη Λαριόχα η παραγωγή μας ε, επεφύλαξαν θερμότατη ε, υποδοχή. Εγώ προσωπικά έλαβα και ε, πρόσκληση να επιστρέψω στη Ριόχα και θα το κάνω, δεν θα διστάσω, είναι πολύ καλή ε, ευκαιρία να επισκεφθώ και πάλι αυτήν την τόσο όμορφη περιοχή. Ευχαριστώ λοιπόν τους διοργανωτές της αποστολής από πλευράς Επιτροπής επίσης, της Γραμματείας Επιτροπής. Σπάνια συμμετέχω στις ημερίδες μελέτης, αλλά πραγματικά ε, εντυπωσιάστηκα Και αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι τα μέλη της γραμματείας άρχισαν να μαθαίνουν και πολωνικά. Ε, νομίζω έτσι ολοκληρώσαμε και το, την μέση διάταξη. Παρακαλώ να έρθετε γέρος για την απογευματινή ε, συνεδρίαση στις 3 η ώρα. Ε, θα υποδεχθούμε τον ε, Έλληνα Υπουργό Γεωργίας. Άρα, μεγαλία. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψή του ε, και θα συζητήσουμε γενικά θέματα καθώς και θέματα χρηματοδότησης. Ζητώ συγγνώμη για τις μικροατέλειες ε, στη, κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας. ζητώ συγγνώμη.